Πριν όμως δώσω το λόγο στον Επίτροπο Στυλιανίδη, τον οποίο χαιρετώ ε, και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας σήμερα το απόγευμα, ε, να πω ότι η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Μογκερίνη, δεν μπορεί να είναι ε, εδώ αυτή τη στιγμή. Να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Στυλιανίδη. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Η Λιβύη βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Η κατάσταση στη χώρα διαρκώς επιδεινώνεται. Ο αριθμός των εσωτερικών εκτοπισθέντων ε, αμάχων έχει αυξηθεί ιδιαίτερα σε περιοχές γύρω από την ε, Μπεγκάζη έχουμε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση σε πολλές περιπτώσεις των υγειονομικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών έχει διαταραχθεί. Πολλά νοσοκομεία και σχολεία μεταβίας λειτουργούν. Η παραγωγή πετρελαίου έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο. Τα αποθέματα σε ρευστό εξαντλούνται και η κυβέρνηση σταματά τη χορήγηση των επιδοτήσεων. Έχει υποβαθμιστεί πολύ τραγικά θα έλεγα το νόμισμα και ε, έχουν ανέβει σε πληθωριστικά επίπεδα οι τιμές για βασικά αγαθά όπως το ψωμί. Η κατάσταση ως προς την ασφάλεια επίσης έχει επιδεινωθεί. Τα μαλαΐ ανακοχές που ε, ορθεσπίζονται σε τοπικό επίπεδο ευπρόσδεκτες βέβαια δεν αρκούν χρειάζεται να επιβληθεί η τάξη και ο νόμος. Πολλές φορές ε, και σε πολλές περιοχές τα διαπρατώμετα έγκληματα μένουν ατιμόρυτα. Συνεχίζεται η λαθρέα διακίνηση μεταναστών από εγκληματικές ομάδες. Τα νότια σύνορα της Λιβύης είναι τελείως αθρά και είναι πολλές οι ζωές εκείνες οι οποίες ε, κινδυνεύουν ε, μέσα στα σκάφη. Όλο και περισσότεροι είναι οι Λίβοι προσπαθούν να ε, φύγουν, να διαφύγουν στο εξωτερικό μέσω της Τινησίας. Με όση βοήθεια και να τους παρέσει, παρέχεται, είναι πολλές οι οικογένειες της Λιβύης οι οποίες έχουν βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση και έχουν εξαντλήσει τους σπόρους τους. Πρέπει να βρούμε μια λύση λοιπόν. Η ένοπλη σύραξη έχει ε, αποβήσει όφελο μόνο ομάδων μαχητών όπω αυτών της ΔΑΕΣ, του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε συνεχιστεί αυτό. Ε, λοιπόν από την ε, συνέχιση του πολέμου και από τα δεινά που αντιμετωπίζει η κοινωνία της Λιβύης. Έχουν οι αρχές προσπαθούν ε, να βρουν ε, κάποια σημεία ε, στήριξης και αν δεν τα καταφέρουν μόνο τους συνεργάζονται με τοπικές πολίτοφυλακές στη Σύρτη, στη Μπεγκάζη και πάλι η κατάσταση είναι δύσκολη και η Ντάες συνεχίζει την επέκτασή του μόνο στη Λιβύη αλλά και σε γειτονικές χώρες. Αυτός είναι λόγος να πιέσουμε για μια κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας που θα εξασφαλίσει και τη θέσπιση των εθνικών θεσμών που χρειάζεται να λειτουργούν. Υπάρχει πρόοδο στην πολιτική διαδικασία. Ο ειδικό απεσταλμένος των Εθνών Μπερναρντίνο Λέονα στον οποίο έχουμε προσφέρει πλήρη υποστήριξη και ενεργό υποστήριξη, κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει την συνεργασία στο Τόμπρουκ της, της κυβέρνησης, της ε, εκλεγμένης κυβέρνησης στο Τόμπρουκ και αντίστοιχα του GNC στο, στην ε, Τρίπολη. Ε, ομόφωνα εξέφρασαν τα Ηνωμένα Έθνη την υποστήριξη στις προσπάθειες του Λέων για το καλό της κοινωνίας των πολιτών. Και είναι καλό να υπογραφούν αυτές οι συμφωνίες όπως προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένες, ε, στην Νέα Υόρκη, στα Ηνωμένα Έθνη. Διαπιστώσαμε μία νέα ελπίδα. Οι γειτονικέ μάλιστα χώρες της Λιβύης, ε, της Λιβύης συμμερίζονται τις θέσεις μας αυτές. Αυτό αποτελεί εν μέρει αποτέλεσμα και των ενεργών πιέσεων που σχέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ώστε να προχωρήσει τόσο πολύ η διαδικασία. Μέρα νύχτα δουλεύαμε κυριολεκτικά για να υποστηρίξουμε την προοπτική μιας κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας. Και τώρα η διεθνής κοινότητα συμφωνεί και παραμένει ενωμένη στο εξής ότι οι Λίβοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να αναλάβουν τώρα την ευθύνη και να σχηματίσουν κυβέρνηση που θα θέσει τέρμα στην κατάρρευση της χώρας. Πολύ καλά γνωρίζουμε ότι ακόμη και αν ε, θεσπιστεί, αν σχηματιστεί η κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας, δεν θα, έρθουν, δεν θα επέλθουν οι αλλαγέ ε, μέσα σε μια μέρα στη Λιβύη. Θα χρειαστεί να περάσει πολλούς χρόνους για να βελτιωθεί η κατάσταση, ακόμη και αν υπογράψουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τη συμφωνία αυτή αλλά πάντως αυτό θα αποτελέσει ευκαιρία για βελτίωση. Δεν θα είναι το, τέλμα, το τέρμα, αλλά η εφετηρία. Και επιτρέψτε μου να εκθέσω τους στρατηγικούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια τις δράσεις που αναλαμβάνουμε και που θα αναλάβουμε προκειμένου να τους επιτύχουμε. Θέλουμε σταθερότητα, ασφάλεια, ε, αξιόπιστη διακυβέρνηση και κράτος δικαίου στη Λιβύη. Ο λαός της Λιβύης αξίζει να ζει σε συνθήκες ειρήνης με ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε να ανθίσει για μια φορά η οικονομία της χώρας και θέλουμε οι λαθροδιακινητές οι οποίοι κερδίζουν από τον πόνο των απεγνωσμένων επιτέλους να ε, χάσουν το πεδίο δράση τους. Πρέπει λοιπόν ε, να εξασφαλίσει τον έλεγχο των συνόρων της η, η Λιβύη και να μπορέσουμε να έχουμε μια νέα κυβέρνηση με την οποία θα μπορούμε να συνεργαστούμε. Αλλά όπως είπαμε και σε όλες τις πλευρές στην Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα πρέπει να ξεκινήσει και ένα πακέτο υποστήριξης 100 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο όμως θα, θα αρχίσει να χορηγείται με το που θα εξευρεθεί η συμφωνία. Σε αυτό προβλέπεται μια σειρά μέτρων χρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα προπολογισμός για τη Λιβύη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθώς και από το μέσο, από το νομοθέτημα συμβάλλουμε στην, Ευρώπη, στην ειρήνη που θα βοηθήσει τους θεσμούς της Λιβύης. Αναλογό μεταξύ, μεταξύ των διαφόρων ομάδων της χώρας θα υποστηρίξει την τοπική διακυβέρνηση, την κοινωνία των πολιτών και βεβαίως και τα μέσα. θα επιτρέψει στους ανθρώπους να ξαναγυρίσουν στην ομαλότητα, στην καθημερινή του ζωή με τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τη δημόσια υγεία. Θα βοηθήσουμε, θα προσφέρουμε βοήθεια σε εκείνα τα Υπουργεία που ασχολούνται κυρίω με τα ζητήματα τη μετανάστευση. Θα βοηθήσουμε τι μικροπεσαίε επιχειρήσει έτσι ώστε να δημιουργηθούν θέσει εργασία, να δοθεί μια ευκαιρία στην νεολαία τη Λιβύη και να επενέλθει στον ορθό δρόμο αυτή η χώρα. Αυτό επιπρόσθετα προς την ανθρωπιστική βοήθεια που ήδη παρέχουμε και η οποία καλύπτει τις πιο επίγουσες ανάγκες των πλέον ευάλωτων ομάδων. Σχεδιάζουμε μια σειρά πρωτοβουλειών για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και για να μπορέσει αυτή η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να γίνει πραγματικότητα. Συνεργαζόμαστε με τα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης, και στο επίγοντα, στο επίγοντα χαρακτήρα προγράμματα, αλλά ε, επίσης και σε πιο μακροπρόθεσμα προγράμματα. Θα θέλαμε να συνεργαστούμε και σε όλες τις, ε, συμμετάσχουμε και σε όλες τις κοινέ ομάδες εργασίας. Ομάδες στην οποία, στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι της διεθνούς κοινότητας και εκπρόσωποι της κυβέρνησης της Λιβύης και οι οποίες συνίστανται αυτή τη στιγμή. Όμως, αυτή τη στιγμή περιμένουμε από τα λιβικά κόμματα να αναλάβουν δράση αποφασιστικά. Κανένας δεν μπορεί να λάβει τις αποφάσεις στη θέση τους ανταυτών. Υπάρχει μεγάλη στήριξη όσον αφορά αυτήν την πολιτική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είμαι σίγουρο ότι θα συνεχίσει να προσπαθεί έτσι ώστε τα εμπλεκόμενα μέρη να βρουν μια λύση, μια σταθερή λύση. Πρέπει τώρα αυτά τα εμπλεκόμενα μέρη να υπογράψουν τη συμφωνία, να αποδείξουν ότι μπορούν να ηγηθούν αυτές τις προσπάθειες για να ξανασταθεί στα πόδια τη Λιβύη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε Στυλιανίδη. Να ξεκινήσει η συζήτηση με τις δηλώσεις από τις πολιτικές ομάδε Από το ΕΛΚ η κυρία Γκάμπριελ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, για την πρώτη φορά από το 2011 έχει ένα φιλοπορία πορεία η Λιβύη για να ολοκληρώσει τη μετάβασή της. Πρέπει να χαιρετήσουμε την εργασία του Μπερναντίνο Λεόν, του ειδικού ε, απεσταλμένου του ΟΗΕ και θα πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά τη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρει παρατηρήσει. Τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του για το καλό του λιβικού λαού, αλλά και για να δοθεί τέρμα σε μια κατάσταση που έχει κάνει αιστεία απειλών για την περιφερειακή ασφάλεια και τη διεθνή τάξη τη χώρα αυτή. Η πίεση διεθνώ πρέπει να διατηρηθεί για να τηρηθούν αυτέ οι υποχρεώσει. Όπω είπατε, κύριε Επίτροπε, δεν υπάρχει χρόνο για την διαπραγμάτευση των όρων, αλλά για την ανάληψη ευθυνών και μόνον. Πρέπει όλοι να αρχίσουν να εργάζονται στο πλαίσιο μια κυβέρνηση εθνική ενότητα. Από την περιφερειακή σκοπιά αλλά και τη σκοπιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπογραμμίσω ότι για όλη την περιοχή του Σαχέλ η γεωγραφική αυτή ζώνη είναι καθοριστική σημασία για να αποφύγουμε την επέκταση τη αστάθεια. Και σωστά αυξάθηκε ο προπολογισμό και τα κονδύλια υποστήριξή μα προ αυτή την περιοχή και την περιοχή του Νίγηρα. Το ίδιο και για το Μαλί. Ε, πρέπει να φροντίσουμε για τη σταθεροποίηση τη κατάσταση στη Λιβύη, όχι μόνο για την αντιμετώπιση τη θερμοκρατία και τη εμπορία ανθρώπων, αλλά και γιατί θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να θυμίσω το έργο τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργασία με του Αφρικανού εταίρου. Υπάρχει ανάγκη από μία ε, κατάρτιση συστήματο ε, ε, συγκέντρωση πληροφοριών για όλη την Αφρικανική Ήπειρο. Και θα πρέπει ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκεντρώσουν τι προσπάθειέ του και να στηρίζουν τι διάφορε πρωτοβουλίε για να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία σε τοπικό επίπεδο με τη συμπερίληψη των γυναικών και των μειονοτήτων. Περισσότερο από ό,τι στη Λιβύη και σε άλλε άλλε χώρε. Χρειάζεται οι γυναίκε να ενισχυθούν για να μπορεί να είναι σταθερή και τοπική εξουσία. Κύριε Επίτροπε, για τη σύγκρουση στη Λιβύη ελπίζουμε να διαδραματίσετε έναν ενεργό ρόλο ε, ενώ όλη η διεθνή κοινότητα ανησυχεί κυρίω για την κατάσταση στη Συρία. Ποιο είναι αυτό το πλεονέκτημα που μπορεί να φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σταθεροποίηση τη ε, ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα υπόλοιπα. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κύριο Μποστινάρο για του σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Ευχαριστώ ε, Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για τις πληροφορίες που μόλις μας δώσατε. Είναι καθοριστική σημασία. Βλέπουμε ότι η Λιβύη είναι από τα μείζωνα θέματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να μα απασχολεί και εδώ. Για την κατάσταση στη Λιβύη, άλλη μια φορά θα επαναλάβουμε αυτό που έχω ξαναπεί. Επανειλημμένο σε αυτό το σώμα. Ε, προθεσμία μετά την προθεσμία. Δεν υπάρχει άλλο χρόνο για χάσιμο. Όμω δυστυχώ κάθε φορά, κάθε μία φορά φαίνεται οι προθεσμίες να παραβιάζονται και η τελική συμφωνία να μην τηρείται. Ούτε συμφωνούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μεταξύ τους. Αυτό δεν μπορεί να είναι πλέον ούτε αστείο ούτε μια αρένα προσωπικών συμφερόντων. Μιλάμε για το πεπρωμένο μιας ολόκληρης χώρας, ενός ολόκληρου λαού και επί της ουσίας για το πεπρωμένο ολόκληρης της Υπήρου. Το μέλλον και η σταθερότητα ολόκληρη τη γεωγραφική αυτή ζώνη είναι αλληλένδετα με το πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Λιβύη. Το ISIS δεν χάνει χρόνο, δεν περιμένει, αλλά απλώνεται και εξαπλώνεται όπου βρει γόνιμο έδαφος. Από εκεί προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει ολόκληρες περιοχές και όχι μόνο μια χώρα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη η διεθνή κοινότητα δεν μπορούν να επιτρέψουν στη Λιβύη να αποτύχει ω κράτο. Θα πρέπει πάνω απ' όλα όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για τη Λιβύη και για του Λίβιου όσοι ε, είναι υπερασπιστέ του να μην επιτρέψουν να αποτύχουν και πάλι ειρηνευτικέ διαπραγματεύσει. Η Λιβύη αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια του λαού τη και των ηγετών τη. Η βία που επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση πρέπει να πάυσει. Όπω ε, ο η εκπρόσωπο έχει πει επανειλημμένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση τίνει χείρα βοηθεία είπε πώ μπορεί να πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία κυβέρνηση εθνική ενότητα στη Λιβύη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει μια συμφωνία να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όλε τι πλευρέ. Όμω, α είμαστε ρεαλιστέ, καμία συμφωνία δεν μπορεί να είναι άψογη για όλε τι πλευρέ τέλεια. Όλοι θα πρέπει να δώσουν κάποια ανταλλάγματα, να κάνουν συμβιβασμού. Και για άλλη μια φορά συζητιέται ένα ειρηνευτικό σχέδιο που έχει προτείνει ο ειδικό απεσταλμένο του ΙΑ και πάλι βλέπουμε μια υπο... επιδείνωση τη κατάσταση. Θα πρέπει να είναι η τελευταία φορά. Στην περίπτωση τη Λιβύη, ο λαό τη χώρα θα πληρώσει το αντίτιμο εάν και αυτή η συμφωνία να βαγίσει. Και μια τελευταία παρατήρηση για αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Να μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση για δύο τουλάχιστον θέματα. Ένα, να σκεφτεί το κατά πόσο πλέον να σε όσους δεν ε, δεχτούν τη συμφωνία και όσους δέχονται την επέκταση των σειράξεων. Ε, ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντέμες Μάκερ για ένα λεπτό. Ε, Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζουμε ότι είπατε εκπρόσωπο και πολύ σωστά αποδίδει την σημασία στην αντιμετώπιση του προβλήματος της Λιβύης. Οι εικόνες που μας έρχονται δεν είναι καθόλου καθησυχαστικές. Είναι αναγκαίο λοιπόν να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των θεσμών στη χώρα, όπως αναφέρατε και εσείς. Μια σειρά από ζητήματα παραμένουν αναπάτητα, όμως δικαιοσύνη, ε, τιμωρία συμφιλίωση, πώς θα εξασφαλίσουμε την συνύπαρξη των διαφορών αυτών ομάδων και φρατριών, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα των εγκληματών πολέμου, πώς θα τιμωρηθούν οι εγκληματίες πολέμου. Οι νέοι θα πρέπει να είναι σε θέση να μάθουν να σκέφτονται μόνοι τους, θα πρέπει να θεσπιστεί μια ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών που θα καλεί τον πολιτικό να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, δώσει απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις, η και η ειρήνη και η σταθερότητα. Δεν θα επιτευχθούν. Πρέπει οπωσδήποτε να δράσουμε και να δράσουμε συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μαούρα Μπαντα... ο κύριος Μαούρα Μπαραντιαράν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, κύριοι συνάδελφοι αυτό το προσχέδιο συμφωνίας που εξετάζουμε σήμερα είναι πραγματικά τελευταία ευκαιρία για τη Λιβύη. Είναι τελευταία ευκαιρία τα εμπλεκόμενα μέρη να ε, δημιουργηθεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας μετά από κατάπαυση του πυρός και να προχωρήσει η χώρα στον δρόμο της ειρήνης. Η χώρα και η περιοχή. Και ιδανικά αυτό θα έπρεπε να γίνει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. 20 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία για να δημιουργηθεί αυτή η κυβέρνηση εθνικής ενότητα. Γιατί διαφορετικά θα ξαναγυρίσουμε στο μηδέν, στην αρχή. Και θα ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσει. Κάτι το οποίο δεν θα είναι μόνο α, τραγικό για τους ανθρώπους τους που ζουν στη Λιβύη, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Θα συνεχίσει η βαλκανοποίηση της χώρας. Θα συνεισφέρει στη δημιουργία και την εμπέδωση του Ισλαμικού κράτους. Αν δούμε τι συμβαίνει στη Συρία και με το ISIS, η Λιβύη μπροστά στο ότι καταφέρνει το ISIS στη Συρία δεν είναι τίποτα. Ε, εάν καταφέρουν ε, να προχωρήσουν, να προελάσουν στην Λιβύη, θα έχουν μετά πρόσβαση και σε πολεμικά πλοία και σε πολεμικά αεροπλάνα σε μια χώρα η οποία βρίσκεται τόσο κοντά στα σύνορά μας και δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε αυτόν τον κίνδυνο. Πρέπει να συνεχιστεί η άσκηση της πίεσης έτσι ώστε τελικά οι διαπραγματεύσεις να τελεσφορήσουν και παράλληλα να παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια προς τις λιβικές αρχές για να καταπολεμήσουν το Ισλαμικό κράτος και να σταματήσουν την προέλασή του. Αυτά είναι τα στοιχεία που θα ε, μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε ένα σταθερό κράτος. Ο κύριος Κούσο Περμού για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται στην ε, Μέση Ανατολή και καλωσορίζουμε τις ε, προσπάθειες στη Συρία και στη Λιβύη. Χρειάζεται μια περιφερειακή λύση στην οποία να έχουν συμμετάσχει όλοι οι ενδιαφερομένοι ε, η Κομισιόν μας μίλησε για τις καταστροφές που συμβαίνουν στην ε, Λιβύη σαν να είναι φυσικές καταστροφές. Να σας θυμίσω κάτι όμως. Το 2011, επί 7 μήνες, οι Ηνωμένε Πολιτείε, το ΝΑΤΟ και οι συμμαχοί του ανέλαβαν στρατιωτική δράση. Η εντολή θεωρητικά ήταν να προστατευθούν οι Λίβοι και να προστατευθούν και οι Ευρωπαίοι. Ακριβώς το αντίθετο συνέβη όμως. Καταστράφηκε η χώρα, καταστράφηκε η Λιβύη, Λιβύη όπως ακριβώς καταστρέφεται τώρα η Συρία. Με εκατοντάδε χιλιάδε χιλιάδες θανάτους αμάχων, εκατοντάδε. χιλιάδες πρόσφυγες και μια περιφερειοποίηση τη σύγκρουση. Η Αφρικανική Ένωση είχε προωθήσει μια συμφωνία, αλλά αγνοήθηκε και αντί αυτή τη συμφωνία από την Αφρικανική Ένωση προτιμήθηκε η ανάληψη στρατηγική δράση. Αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη γίνονται επαφέ για να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση εθνική ενότητα. Αυτό πραγματικά χρειάζεται να οδηγήσει τελικά στη δημιουργία μια τέτοια κυβέρνηση, αλλά για να συμβεί θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα πολιτικά κόμματα, όλε οι πολιτικέ φωνέ, για να μην ε, καταλήξουμε σε μονομερή στρατηγική δράση. Ευχαριστούμε για 1,5 λεπτό, κυρία Λοκμπίλερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Μόλις επιστρέφω από την, από την Τίνιδα, όπου είχα συνομιλίες ε, και με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, ε, ακτιβιστών και άλλων της ε, Λιβύης. Πολιτική ενότητα λοιπόν είναι μια ιδέα την οποία υποστηρίζουν. Αλλά καταγγέλνουν ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη ηγετικών μορφών. Είναι θετική η συμβολή Τη προτάσεω για την προστασία των εθνικών δικαιωμάτων και κυρίω την τιμώρηση των εγκλημάτων. Αλλά δεν μπορούμε και να απαυκαλιζόμαστε. Η εξάσφυλληση μια συμφωνία είναι πολύ σημαντική, αλλά και πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχει πληθώρα φυλακών που επιδιώκουν διαφορετικά συμφέροντα η κάθε μία και δεν πρόκειται όλε να υπογράψουν. Και μία λοιπόν να μην υπογράψει. Υπάρχει ο κίνδυνο τη κλιμάκωση τη βία. Ε, είναι όλο και πιο δύσκολη η κατάσταση οικονομικά και, και κοινωνικά. Υπό τι συνθήκε αυτές η δημιουργία μιας, ε, μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας είναι τεράστια πρόκληση και θα χρειαστεί περισσότερη και μεγαλύτερη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό, εάν ε, μιλήσουν τα κράτη-μέλη με μία και μόνο φωνή, θα καταστεί ακόμη πιο αποτελεσματικό. Έχουμε δει φρικτές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Λιβύη, σφάρος Λιβύων πολιτών ε, ή προσφύγων. Πιστεύω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να υποστηρίζει τις ε, προσπάθειες των αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα και έξω από τη Λιβύη και να συμβάλλει στο δυνατόν στην ειρηνευτική διαδικασία. Ευχαριστούμε ο κύριος Καστάλντο για ένα μισή λεπτό και εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αφού γίνει συμφωνία θα πρέπει πάνω απ' όλα να πείσουμε τα μέλη που έχουν συμβληθεί. Αυτή η φράση του Καβούρ νομίζω ότι μπορεί να ισχύσει και για την τωρινή κατάσταση στη Λιβύη. Νομίζω ότι πρέπει να χαιρετήσουμε το έργο του Μπερναντίνο Λεόν για μια κυβέρνηση εθνική ενότητα και ακόμα και αν δεν έχει επιτύχει το σχέδιο, πρέπει να ξέρουμε πώ αντιστέκονται οι φυλέ στα νότια τη χώρα και αλλού. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει προσπάθεια για τον έλεγχο των νότων σύνορων τη χώρα. Ελπίζουμε η δράση μα να μην φτάσει πολύ αργά και να μην οδηγήσουμε τη χώρα και σε άλλο εμφύλιο πόλεμο. Σε κάθε περίπτωση, οι αλχημίε του σχεδίου του ΟΗΕ δεν φαίνεται να έχουν φέρει την επιθυμητή λύση. Και βεβαίω υπάρχει στρατιωτική ε, κλιμάκωση, κλιμάκωση των σειράξεων στη Βεγγάζη. Αλλά και στο Τομπρούκ με τη στρατιωτική κυβέρνηση ε, υπάρχει αντιπαράθεση με, το, ε, με την κυβέρνηση τη Τρίπολη. Πρέπει λοιπόν, ενώ η Πρωθυπουργή του Μαρόκου, του Μαρόκου προειδοποιεί να ε, σκεφτούμε ότι δεν έχει φτάσει η ώρα της ειρήνης και της σταθεροποίησης. Το μέα κούλπα του Προέδρου Ομπάμα τον Σεπτέμβριο στο ΝΟΙΕ που ε, μετανιώνει για τα ασφάλματα του παρελθόντος δεν μου φέρεται ούτε καν ε, αξιόπιστο σε τοποθέτηση. Μου φαίνεται υποκριτική στάση όπως και της κυβέρνησης Μπούς. Στην πραγματικότητα οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία είναι οι μεγάλε δυνάμει που με ελαφρότητα οδήγησαν σε διάλυση τη χώρα χωρί να ανησυχήσουν για τη δημοκρατική τη μετάβαση. Οι ορέξει του για το πετρέλαιο τη Λιβύη ήταν πιο σημαντικό από την ειρήνη που θα πρέπει να επικρατεί στη χώρα. Τι ευθύνε λοιπόν αυτέ, λέγατε επίτροπε, πρέπει να τι αναλάβουμε. Συμφωνώ, αλλά πότε οι υπεύθυνοι αυτή τη καταστροφή θα αναλάβουν τι δικέ του. Κύριε Καστάλντο, καλά για κάρτα για σα. Ναι. Τη δέχεστε. Από τον κύριο Γιάκοφτσιτ. Παρακαλώ. Κύριε Ευρωβουλευτέ, ευχαριστώ καταρχήν που δεχτήκατε την μπλε κάρτα μου. Συμφωνώ απόλυτα. Μήπω Μήπως μπορείτε να επαναλάβετε κύριε Γιακόφτσιτ. Δεν είναι δίκαιο να, το, την υποβάλω στα Ιταλικά την ερώτηση. Θα μιλήσω κρατικά. Ευχαριστώ λοιπόν που δεχτήκατε την μπλε κάρτα μου και θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την ανάλυση σας για την κατάσταση και την διάλυση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Λιβύη. Ε, όμως ε, κάποιοι αναλυτές λένε ότι για τη λύση στη Λιβύη και στη Συρία θα πρέπει να υπολογίζουμε στη Βοσνία Ριζαγοβίνη. Ε, να παραδειγματιστούμε από αυτή. Σα διαβεβαιώ όμω ότι δεν λειτουργεί καθόλου το κράτο στη Βοσνία Ερζεγοβίνη παρά την ειρήνη που υπάρχει. Συμφωνείτε λοιπόν ότι θα πρέπει πρώτα να αφήσουμε του λαού ε, τη Λιβύη και τη Συρία από μόνοι του να λύσουν το πρόβλημα και εμεί απλώ θα του διευκολύνουμε να πάρουν εκείνη τα χέρια το πεπρωμένο του. Ευχαριστώ συνάδελφε Γιάκοπτη. Συμφωνώ απολύτω μαζί σα όπως και οι συμφωνίε στην Τετώνα έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές, είναι καλές για μια προσωρινή είναι για μια εκεχηρία. Όμως δεν μπορούν να οδηγήσουν σε καλή διαχείριση την κρατική δομή ενός κράτους. Θα πρέπει λοιπόν να μην διαπράξουμε τα ίδια σφάλματα και να μην ε, περάσουμε στα ίδια μεγάλα λάθη. Διότι πάλι θα οδηγηθούμε σε παράλυση και θα έχουμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα να λύσουμε μετά από λίγα χρόνια η κυβέρνηση δεν έχει αποτελεσματική, ε, αποδειχθεί αποτελεσματική για να αντιμετωπίσει τη δράση του ΆΙΖΙΣ. Ευχαριστούμε ο κύριος Μποργκέτσο για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Περίπου 10 λεπτά μίλησε ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Και μας παρουσίασε και εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ε, θέση της και την άποψή της. Και ζητώ συγγνώμη, αλλά βλέπω ότι παρά την παρουσίαση που μας έκανε τη κατάσταση, είπατε εκπρόσωπος δεν κατέληξε σε κανένα συμπέρασμα. Ούτε εκπρόσωπος επιτροπή. Οπότε δεν καταλαβαίνω τελικά. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο συγκεχημένη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λιβύη, που είναι μια γειτονική χώρα τη Μεσογείου. Η κατάσταση είναι κατεπίγουσα. Η ανάγκη επιτακτική ε, να καταπολεμηθούν οι μαφίες ε, των διακινητών και των δουλεμπόρων. Η κατάσταση στη Λιβύη είναι απελπιστική και η δήλωση του Δίλα Αλγαριάνη, του μεγάλου μουφτή, τι έλεγε. Ότι ο Ισλαμικός νόμος, η Σαρία, είναι το μέλλον στη και αυτή θα είναι η μοναδική πηγή δικαίου. Και η Σαρία θα είναι ο μοναδικός νόμος που θα ισχύει στη Λιβύη. Αυτά είπε ο Μέγας Μοφτής. Τι γνώμη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη νέα κατάσταση της ε, εθνικής ενότητας ε, που υποτίθεται ότι προωθεί ο Οργανισμός Εθνών γιατί οι Ευρωπαίοι λάμουν της απουσίας τους. Τελικά η Σαρία θα είναι το μέλλον για τη Λιβύη. Ο κύριος Επιτίδιος για ένα λεπτό. Η περίπτωση της Λιβύης είναι μία ακόμη απόδειξη της ασφαλμένης εξωτερικής πολιτικής που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενεπλάκη, χωρίς να υπάρχει λόγος και κυρίως χωρίς να εξυπηρετούνται τα συμφέροντά της, στον πρώτο από τους δύο εμφυλίους πολέμους της χώρας με αποτέλεσμα αντί να επιλύσει το πρόβλημα να κατορθώσει να γίνει μέρος του προβλήματος. δημιουργήθηκε ανθρωπιστική κρίση όλες οι ενδυναμωνόμενες παρατάξεις παραβίασαν και εξακολουθούν να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και κύματα προσφύγων ετούντων άσυλο ε, και μεταναστών οδηγήθηκαν στην ευρώπη μέσω της ιταλίας. ακόμη χειρότερα στη χώρα αναπτύχθηκαν ισχυρέ δυνάμει των τζιχαντιστών του isis. κάτι ανάλογο συνέβη και με τη συρία. Η σπίσμα της εξελίξεως των γεγονότων άρα και της λογικής η ευρωπαϊκή ένωση εξακολουθούσε να επιμένει στην ανατροπή του προέδρου ασαντ. τα αποτελέσματα τα γνωρίζετε. ομοίως και με την τουρκία. η ευρωπαϊκή ένωση ανέχθηκε την τουρκία να υποστηρίζει τις δυνάμεις του isis και να προωθεί χιλιάδες παράνομους μετανάστες στην ελλάδα και μέσω αυτής στην ευρώπη. και τώρα τι κάνει η ευρωπαϊκή ένωση ζητά από την τουρκία να κάνει το αυτονόητο και την αναδεικνύει σε προνομιούχο συνομιλητή αντί να τη υπενθυμίζει ότι είναι χώρα προ ένταξη και οφείλει να είναι συνεπή στι υποχρεώσει τη. εάν λοιπόν δεν απαλλαγούμε από τι αιμονέ στην εξωτερική μα πολιτική δεν θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα απλώ θα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματά του. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι τέσσερα χρόνια σοβεί εμφύλιος πόλεμος στη Λιβύη. Αυτό έχει τελείως καταστρέψει τη χώρα και ε, όλους τους θεσμούς της τους όποιους θεσμούς με το παλιό καθεστώς. Και σήμερα επικρατεί πλήρες χάος. Ένα ε, χάος που αποτελεί κίνδυνο για την περιφερειακή σταθερότητα, αλλά και τη ε, σταθερότητα της Ένωσης είναι πλέον ένας χώρος όπου οριάζουν τα λαθρεμπόρια, η λαθρομετανάστευση και βέβαια φυσικά προς τις χώρες μας. Έρχεται εδώ να προσθεθεί και ε, η τρομοκρατική απειλή. Ε, έχει εγκατασταθεί το Ισλαμικό κράτος στη Λιβύη και είδαμε τι συνέπειες έχει αυτό για την γειτονική χώρα την Ισία, όπου ε, οι τρομοκρατικές επιθέσεις έγιναν ε, ε, από άτομα που προέρχονται από τα λιβικά τρομοκρατικά δίκτυα. Χαιρετίζω τις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τερματίσει την ε, κρίση στη Λιβύη και υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών έχουμε τώρα την επιχείρηση Σοφία, αλλά για να στεφθεί με επιτυχία αυτό θα γίνει μόνο εφόσον η Λιβύη έχει σταθερή κυβέρνηση ε, εθνικής Ενότητας, συνομιλητή της Ένωσης. Ο Μπερναντίνο Λεόν έχει διαπραγματευτεί ένα κείμενο που είναι η συμφωνία της τελευταίας ευκαιρίας. Τρεις ε, απόπειρες ε, υπογραφής μιας συμφωνίας να βάγισαν. Στις 20 Οκτωβρίου τώρα έχουμε μια καταληκτική ημερομηνία και δεν θα ήταν καθόλου ενθαρρυντικό μήνυμα να ζητήσει παράταση το Λιβικό ε, Κοινοβούλιο. Το Λιβικό Κοινοβούλιο. Ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να ε, προχωρήσει και να εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Έχετε μία μπλε κάρτα. Τη δέχεστε από πλευράς του κυρίου Σοπχάντα. Σας παρακαλώ. Εάν δέχεστε φυσικά κύριε Πρέντα να απαντήσετε. Όχι. Εγώ δεν συζητώ με το εθνικό μέτωπο. Μάλιστα. Ο κύριος Παντσέρη, για 1,5 λεπτό. Grazie. Ευχαριστώ. Grazie. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βρισκόμαστε στη πιο περίπλοκη φάση τώρα ε, θα πρέπει όλοι να έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος. Είναι απολύτως απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει όλη την απαραίτητη πίεση έτσι ώστε να προχωρήσει μια συμφωνία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων στη Λιβύη και μάλιστα πριν την 20 Οκτωβρίου. Ε, δεν θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω ολιγορίες και ε, καθυστερήσεις. Είναι δύσκολη πάντα η τελική ευθεία, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν οι πάντες ότι έχουν ευθύνη. Διότι ε, αυτοί που δεν θα αρθούν στο ύψος των ε, περιστάσεων θα έρθουν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους στο μέλλον. Νομίζω ότι δεν ήταν καλή ιδέα αυτό που ακούσαμε τώρα για την κατάσταση του Μπεραρδίνο Λεόν. Ε, είναι κακή ιδέα αυτή. Θα πρέπει να τον βοηθήσουμε στην τελική φάση και όχι να τον αντικαταστήσουμε για να φτάσουμε σε τελική συμφωνία. Αλλιώς θα αυξηθούν τα προβλήματα και στην περιφέρεια και στην Ευρώπη. Διότι θα μπορούσε ε, διαφορετικά να επεκταθεί η αστάθεια, η τρομοκρατία. Είναι χιλιάδες ε, οι εκτοπισμένοι στα ε, σύνορα Λιβύης την Ισίας, με ό,τι αυτό σημαίνει και με τη διακίνηση ανθρώπων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί συμφωνία, ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ό,τι περνάει από τα χέρια της για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Είναι πάρα πολύ λίγες ημέρες που μένουν και θα πρέπει να βιαστούμε. Έχετε ερώτηση από τον κύριο Κάρβερ. Τη δέχεστε, μπλε κάρτα. Παρακαλώ, κάντε την ερώτησή σας κύριε Κάρβερ. Ευχαριστώ κύριε Παντσέρη. Πολύ επικριτικός ακούγεστε για τα Ηνωμένα Έθνη. και με κάπως αλαζονικό τρόπο λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, εκείνος ο διεθνής οργανισμός που θα λύσει το πρόβλημα. Είστε τόσο βέβαιος, έχει πια τόσο λαμπρές επιδόσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μην εμπιστεύεστε τα Ηνωμένα Έθνη. Μήπως πρέπει να δείτε τη συνολικότερη εικόνα γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Απάντηση. Νομίζω ότι δεν καταλάβατε πάρα πολύ καλά τα όσα είπα εγώ. Εγώ δεν επέκρινα ούτε τα Ηνωμένα Έθνη ε, για τη δράση τους ούτε τίποτα. Είπα ότι είναι λάθος η αντικατάσταση αυτή τη στιγμή του Μπερναρντίνο Λεόν. Δεν θα έπρεπε να ανοίξει τώρα αυτό το θέμα. Δεν είναι του παρόντος διότι έτσι ε, αποδυναμώνεται ο διαπραγματευτής. Γι' αυτό μόνο επέκνα τον ΟΗΕ. Η σημερινή καταστροφική κατάσταση στη Λιβύη είναι από τις σημαντικότερες ήττες της παγκόσμιας πολιτικής και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής ε, τις τελευταίες δεκαετίες. Ε, δείχνει την υποκρισία των ελίτ της δύση. γιατί στην εποχή του Καντάφη συνεργαζόταν μαζί τους λόγω του πετρελαίου ουσιαστικά υποστηρίζοντας ε, τους τρομοκράτες ε, και ε, πολλοί φωτογραφίζονταν ε, οι ηγέτε της Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Καντάφη. Τώρα έχουμε με ένα τελείω διαφορετικό σενάριο. Οι χώρες χώρε που συνεργάζονται με τον Καντάφη συνεχίζουν να επιδιώκουν τα αμυγό οικονομικά του συμφέροντα και υπό το πρόσχημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέτρεψαν τον Καντάφη και τώρα ζητούν την ελληνική από όλες τις χώρες για να επιληθεί η προσφυγική κρίση. Η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία που δεν είχαν καμία σχέση με το καθεστώς του Καντάφη ε, βρέθηκαν στην γενική κατακραβή ε, γιατί δεν ε, θέλουν να αναλάβουν την συνυπευθυνότητα για την κρίση στην Αφρική. Η μυρωδιά του πετρελαίου της Λιβύης που δελέασε πολλές χώρες της Δύσης δεν τους δίνει καμία ε, ηθική υπεροχή για να δίνουν μαθήματα σε άλλες χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Έτεριτς θέλει κύριε Κάσκη να σας υποβάλει μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Κάντε την ερώτησή σας κύριε Έτεριτς. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που δεχτήκατε την ερώτηση κύριε Κάσκη. Συμφωνώ εν γέννη με αυτά που είπατε. Συμφωνείτε ότι είναι ηρωνία να έχουμε χώρες ε, όπως ε, το Ηνωμένο Βασίλειο που επί Μπλερ ε, φλέρταρε με τον Καντάφη και άλλες χώρες τάχθηκαν κατά της Λιβύης. Θεωρείτε ότι είναι ηρωνία ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι μπορούν να λύσουν τα προβλήματα, ενώ αυτοί ουσιαστικά ήταν οι και προκάλεσαν όλα αυτά τα προβλήματα. Συμφωνείτε μαζί μου. Κάσκιο. Σε ό,τι αφορά τους ηγέτες ε, κάποιο χώρο εγώ σκεφτόμουν περισσότερο τους ηγέτες ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Ο κύριος Νάρτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξή. Καταρχήν δεν υπάρχει Λιβύη. Δηλαδή δύο βουλές οι οποίες δεν εκπροσωπούν κανέναν και δύο κυβερνήσει που δεν κυβερνούν. Αυτό που έχουμε είναι φυλές είναι ομάδες, είναι ε, ιδιωτικοί στρατοί, οι οποίοι απλώς προσπαθούν να κερδίσουν ε, εδάφη ε, και επιρροή στα διάφορα λαθρεμπόρια. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία μαύρη τρύπα, η οποία αποτελεί αρχή τέλος και σημείο διέλευσης για όλα τα επικίνδυνα λαθρεμπόρια είτε σε ανθρώπους, είτε σε ναρκωτικά, είτε σε όπλα. Έχουμε επίσης και το ISIS το οποίο ενώνει ως κομβικό σημείο όλα τα παραπάνω που δημιούργησε μια κυβέρνηση που δεν θα κυβερνήσει αλλά που θα διεκδικεί με κάποια προφανή νομιμότητα την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας. Δηλαδή στρατιωτική επέμβαση από τη Δύση ε, έτσι ώστε οι αντίπαλοι να εξοδοθούν. Αυτά λέμε σε συμφωνίες στη Νέα Υόρκη και πρέπει να σας πω πως δυστυχώς υπό αυτές τις φρικτές συνθήκες θα πρέπει εμείς να στηρίξουμε αυτή τη φαντασίωση ε, του Μπερναρδίνου Λεόν, γιατί πρόκειται περί απλής φαντασίωσης. Un minuto anche per lei. Ο κύριος Βαλέ, η κυρία συγγνώμη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη έχασε ε, γιατί ουσιαστικά πήγε, ανέτρεψε τον κατάφυγο, βάρδισε και έφυγε χωρίς να έχει ένα σχέδιο τι θα γίνει με τη Λιβύη και ποια θα είναι η μοίρα της μετά την ανατροπή του Καντάφη, πώς θα δημιουργηθούν ε, κρατικές δομές. Ε, και η Λιβύη έγινε κόμβος ε, λαθρεμπορίου όπλων. Είχαμε συνάντηση με εκπροσώπους των αρχών της Τινησίας και της Λιβύης και μας είπαν ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί το νέο σχέδιο η επιχείρηση Σοφία. Κανένας δεν μας είπε ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανασφάλεια και σε έλλειψη της ε, προστασίας του λιβικού λαού. Φαίνεται όμως είναι ε, ένα θέμα πολύ σημαντικό. Παρόλο που εμείς θέλουμε να σταματήσουμε το προσφυγικό κύμα, δεν νομίζω ότι έτσι θα βοηθήσουμε το λαό της Λιβύης. Κύριος Χούκερ. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί νομίζει, είπατε εκπρόσωπος, πως θα επηρεάσει την πολιτική σκηνή στη Λιβύη. Γιατί θα δημιουργηθεί αυτή η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας όταν δεν υπάρχει ενότητα. Ούτε στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε τι γίνεται με το πώς αντέδρασαν οι διάφορες χώρες στην τρέχουσα κρίση με τη μετανάστευση. Ξέρετε τι συνέβη μετά την παρέμβαση της στη Λιβύη. Ξέρετε πώς ήταν η συλλογική αποτυχία των χωρών μας έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ειρήνη στην ε, Βόρειο Αφρική. Ξέρετε ποιο είναι το κενό εξουσία στη Λιβύη. Ο πρόεδρος Ομπάμα υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει πως αποτύχαμε και δημιουργήσαμε ένα χώρο ανάπτυξης τρομοκρατών του Ισλάμ, όπως για παράδειγμα το ISIS, που έχουν δημιουργήσει εγκληματικές αυτοκρατορίες ε, μέσα σε αυτό τον, που έχουν καταφέρει να διεισδύσει στον ίδιο τον ιστό ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τον έχουν πλημμυρίσει με τους δικούς τους μαχητές. Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα του πόσο έχει αποτύχει η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια και η σωματεμπορία και το λαθρεμπόριο ανθρώπων από τη Λιβύη έχουν δημιουργήσει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να προσπαθεί την κρίση μετανάστευση να τη λύσει μια και έξω, ζητάνε περισσότερη κεντρική διαχείριση του προβλήματος με μια ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή ευρωπαϊκή. Δηλαδή, δεδομένου του ότι έγινε με την ευρωπαϊκή διαχείριση του ευρώ, εγώ δεν θα εμπιστευόμουν μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή για να εξασφαλίσει τα δικά μας σύνορα και τις ε, ακτές και για να μας δώσει μαθήματα ευρωπαϊκής διαχείρισης της πολιτικής μας. Σας παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο, γιατί διαφορετικά θα παρατείνουμε υπερβολικά τη συζήτηση. Ο κύριος Σοπράντα έχει το λόγο. Από το 2014 η Λιβύη είναι η άμεση συνέπεια της ε, ε, επέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011 και είναι ένα αποσαθρωμένο, διαρρεμένο κράτος, διαλυμένο με δύο κοινοβούλια, δύο κυβερνήσεις και δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις. Η Τρίπολη στη Δύση με ισλαμιστική κυβέρνηση στηρίζεται σε μια κυβέρνηση που δεν έχει αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη και σε ένα στρατιωτικό συνασπισμό που τη στηρίζεται από την Τουρκία και την Κατάρ. Ε, ανατολικά έχουμε την κυβέρνηση του Τομπρούκ με πρώην καταβιστές φεντεραλιστέ που αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, τη Σαουδική Αραβία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, και στηρίζεται στο στρατιωτικό συνασπισμό του στρατηγού Χαφτάρα ε, κατά των ε, Ισλαμιστών της Βενγάζης. Οι Ισλαμιστέ συνεργάζονται με τους Σιχαϊστές του Ισλαμικού Μαγκρέπ, της Αλκάιντα και άλλων και με την Αίγυπτο που έχουν και ένα βάση επιπλέον αυτού του Σινά χωρίς να ξεχνούμε την, τις δράσεις του Ισλαμικού κράτους το 2014. Επίσης την Κυριναϊκή σε μια επαρχία που δίνει ε, στρατηγικό πλονέκτημα στο Ισλαμικό Χαλιφάτο έχει και πρόσβαση στη θάλασσα. Και σήμερα για να προστατεύσουμε την Ευρώπη μία μόνο υπάρχει ένα ε, ναυτικό αποκλεισμό των ε, λιβικών ακτών για να σταματήσουμε στην πηγή την, ε, των απόπλου πλοίων που γεμάτα πρόσφυγες στέλνονται από διακινητές και πολλές φορές να βαγούν και στη Μεσόγειο. Μακρηγορήσατε. Ο κύριος Γκόλνης, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας τον συνάδελφο Σοπράντ έχω την αίσθηση ε, ότι ακούω το Θωμά τον Ακινάτη. Ε, διαρριγνύει τα ημάτια του και ε, περιγράφει πολύ καλά την κατάσταση. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλει ο κ. να συζητήσει μαζί μας, γιατί οι πολιτικοί του φίλοι ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση. Να, τους, ονομάσουμε. Ο κ. Καντάφη ε, υπό την έμπνευση του κυρίου Μπερνάρα Ρίλεφη, ο οποίος τον καλοδέχτηκε και τον άφησε να στήσει και τη σκηνή του κοντά στο Ελίσια Παιδεία με 100 μέτρα κόκκινο χαλί και αφού ε, ε, τον εναγκαλίστηκαν με πρώτη ευκαιρία τον μαχαίρωσαν πισόπλατα και συμμετείχαν και στη δολοφονία του. Ε, τουλάχιστον αυτό ας μας γίνει μάθημα. Να μην αποσταθεροποιήσουμε εμείς η Δυτική και, και άλλη χώρα. Το Ιράκ αποσταθεροποιήσαμε και τη Λιβύη και ετοιμαζόμαστε τουλάχιστον ορισμένοι εδώ μέσα να αποσταθεροποιήσουν και τη Συριακή κυβέρνηση. Αυτή είναι η πολιτική που ανοίγει το δρόμο για τους εξτρεμιστές, τους Ισλαμιστές και που κατά τα άλλα υποτίθεται ότι καταπολεμάται. Ο κύριος Γκάλερ για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι το καλύτερο που μπορεί κανείς να διαπιστώσει σήμερα είναι το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα γενικά υποστηρίζει το σχέδιο του Μπερναντίνο Λεόν. Καλό είναι αυτό από μόνο του, αλλά δεν μας βοηθάει δυστυχώς την κατάσταση που σήμερα έχουμε περιέλθει και καλό είναι ε, για την περίπτωση πολιτικής συμφωνίας να είμαστε έτοιμοι και με ένα υποστηρικτικό πακέτο. Αλλά φοβούμε ότι δεν πρόκειται να το καταφέρουμε το επόμενο διάστημα αυτό. Όπως ακούμε, ε, τόσο και ε, η πλευρά της Τριπόλεως δεν υποστηρίζεται πια από το Μαρόκο, το οποίο έχει σταματήσει, αλλά και από ό,τι φαίνεται και ε, ε, η Βουλή στο Τομπρούκ έχει διευρύνει την εντολή της για το διάστημα μετά τις 20 Οκτωβρίου. Άρα ε, είναι μάλλον ζωφερή η κατάσταση και καθόλου ρόδινες οι Υπάρχουν και πολιτοφυλακές που δεν έχουν κανένα συμφέρον στην Τρίπολη και στο Τομπρούκ να συμφωνήσουν γιατί κάνουν εκεί τις εγκληματικές τους δραστηριότητες και διάφορες άλλες business. Υπάρχουν όμως ε, και άλλες δυνάμεις διαφορετικές που υποστηρίζουν την Τρίπολη και το Τομπρούκ. Ε, το Τομπρούκ είναι η αναγνωρισμένη νόμιμη κυβέρνηση, αλλά ποιος υποστηρίζει την Τρίπολη. Το Κατάρ λέει η Τουρκία και το Σουδάν. Και για μένα τίθεται το εξή ερώτημα. Με την Τουρκία έχουμε έτσι και αλλιώς συνομιλίες. Δεν θα μπορούσαμε εκεί να ρωτήσουμε τι συμφέροντα μπορεί να έχει η Τουρκία ε, τα οποία εξυπηρετεί η κυβέρνηση της Τρυπόλεως και δεν είναι σε θέση ούτε πρόθυμη να ε, βοηθήσει για να βρεθεί λύση. Νομίζω θα ήταν χρήσιμο αυτό και σημαντικό να το θέσουμε υπόψη των Τούρκων στις συνομιλίες που έχουμε μαζί τους. κυρία κυρία Γκόμες, μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Τι να πούμε για το χάος και την ανθρωπιστική καταστροφή στη Λιβύη. Εμείς βοηθήσαμε να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση εξαιτία έλλειψης συντονισμού και ασυνεννοησίας ε, και δεν συντονίσαμε την ευρωπαϊκή δράση μετά την ανατροπή του Καντάφη. Και έτσι ουσιαστικά αφήσαμε τους παραστατητικούς να μετατραπούν σε ε, τρομοκρατικέ τρομοκρατικές συμμορίες. Και μάλιστα η συμφωνία που προτείνει ο ΙΕ δεν πρόκειται μάλλον να υπογραφεί σύντομα με βάση αυτά που ακούμε από το, το και την Τρίπολη. Και μάλιστα η καταστροφή στην Ιεμένη φαίνεται ότι είναι ε, ε, προετοιμασία και ενέργεια του Χαφτάρ ε, που υπολογίζεται στις αλαφίτες μαχητές. Και αυτές, αυτό θα έχει τρομοκρατικές συνέπειες για το λαό της Λιβύης και τους ξένους που προσπαθούν να φύγουν όπως όπως και να καταλήψουν τη χώρα. Η αποτυχία δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλεται στην έλλειψη ενότητας και την αντιπαράθεση και την αντιδικία μεταξύ των κρατών μελών για τα για το πετρέλαιο και άλλα συμφέροντα. Γι' αυτό κάποιε ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε είναι πολύ πιο εκτεθειμένε απέναντι στη, Συρβή, στη Λιβύη και μάλιστα σκέφτονται και στρατιωτική επέμβαση με αποστολή στρατευμάτων ξηρά. Ε, πολύ δύσκολο βέβαια να βρουν αμοιοποίηση για κάτι τέτοιο. Ε, κανένας δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι όλα οφείλονται στις, ε, στην εσωτερική αντιπαράθεση των φατριών και να μην ξεχνούμε τον πόλεμο δι' αντιπροσώπου που γίνεται στη Λιβύη, τη Σαουδική Αραβία ε, ε, και, των Σαουδικό, και των Ηνωμένων ε, Εμμυράτων στο Τομπρούκ και του Κατάρ και τη Τουρκία μέσω τη Ισλαμική Αδερφότητα στη Μισράτα. Αν δεν σταματήσουμε αυτό τον πόλεμο δι' αντιπροσώπου, δεν θα μπορέσουμε να παρεμποδίσουμε την επέλαση του Νταές του Ισλαμικού κράτους και στη Λιβύη και ουσιαστικά θα στραφούμε και κατά του ευρωπαϊκού λαού. Κύριο Μπέλντερ, για ένα λεπτό, ευχαριστώ πρόεδρε. Η χώρα των πολιτοφυλακών είναι η Λιβύη. Και αυτό το καιρό ε, ζει ένα εμφύλιο πόλεμο με δύο παράλληλες κυβερνήσεις και δύο παράλληλες βουλές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπα ε, ότι εκπρόσωπος θα ήθελα να μου απαντήσει ή μάλλον θα μου απαντήσει γραπτός. Ε, κινδυνεύει η Ευρώπη ισχύουν αυτά που ακούμε ότι οι Τούρκοι στέλνουν ε, όπλα εκεί στους Λίβιους Ισλαμιστές και αν ναι το έχουμε θέσει αυτό υπόψη της Τουρκίας το είπε και ο κύριος Γκάλερ έχω την ίδια ερώτηση δεύτερον ποια θέση παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε σχέση με παραδόσεις όπλων από τη Ρωσία προς την κυβέρνηση του Μπρουκ την οποία κατά τα άλλα αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τις απειλές του Ισλαμικού κράτους στη Λιβύη που είναι οι τεράστιες ροές ε, προσφύγων και μεταναστών. Τα έχουμε λάβει αυτά υπόψη μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάουτμανς για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή. Νομίζω πραγματικά ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη και το είπαν πάρα πολλοί συνάδελφοι ήδη. 400.000 άνθρωποι εντό της Λιβύη έχουν τραπεί σε φυγή και τόσο, τόσοι πολλοί άλλοι ψάχνουν ε, τη σωτηρία τους και ε, κινδυνεύει να γίνει υγρός τάφος η Μεσόγειος για εκατοντάδες χιλιάδες. Εμείς εκκλήσεις κάνουμε, αλλά έχει έρθει η ώρα να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές και ε, γι' αυτό χρειάζονται την υποστήριξή μας οι Λίβοι. 100 εκατομμύρια νομίζω έχει ε, έτοιμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει ε, τη δημοκρατική ε, μετάβαση της χώρας. Είναι καλό αυτό, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται βοήθεια, όχι μόνο χρηματική, επιτόπου, με τα Ηνωμένα Έθνη, με γνώση, με τεχνική υποστήριξη, αστυνομίας, δικαιοσύνης. Θα πρέπει να τολμήσουμε να μιλήσουμε για ξανά ε, συνεργασία που έχει διακοπεί για την αστυνομία και το στρατό. Και ένα τελευταίο, ε, θα ήθελα να μιλήσω για αυτό ε, που Rights Watch να προσαχθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρούσικ. Αν δεν ανάψετε το μικρόφωνο σας κύριε Μαρούσικ δεν πρόκειται να σας ακούσει κανείς. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι το πρώτο θύμα κάθε πολέμου είναι η αλήθεια. Ε, γιατί αν μας ε, λείπει η αλήθεια, ε, γινόμαστε θύματα της προπαγάνδας και του λακισμού και της δημαγωγίας. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το πρόβλημα να λύσουμε, της αλήθειας. Η Ευρώπη είναι άρρωστη. Και δυστυχώς ε, δεν αρκεί να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα της αρρώστιας, αλλά τα αίτια της. Και τα αίτια της αρρώστιας είναι άγνωστα. Η Λιβύη, όπως και άλλες χώρες της ε, Βόρειας Αφρικής ή της Ασίας, ε, καταστράφηκε με συμμετοχή των δυτικών δυνάμεων. Έτσι καταστράφηκε το Ιράκ. Και δημιουργήθηκαν πολλές ερμηνείες και μας δίνονται πολλές εσφαλμένες ερμηνείες. Το ίδιο γίνεται και στην Λιβύη, γιατί ε, συγκαλύπτουμε την αλήθεια για τα αίτια του κακού. Και όταν εθελοτυφλούμε για την αλήθεια δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Θα πρέπει να μας πούνε οι δυτικές κυβερνήσεις ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες για το ότι βυθίζεται η Ευρώπη. Για να ξέρουμε γιατί βυθιζόμαστε, γιατί καταστρεφόμαστε. Αυτή πραγματικά είναι η τραγωδία καταστροφή της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Ο κύριος Μπαλτσό, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το 2011, στα πλαίσια της Αραβικής Άνοιξης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισαν ότι και στη Λιβύη θα πρέπει αμέσως να επικρατήσει η δημοκρατία. Και με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ ανέτρεψαν τον τότε δικτάτορα. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι ακριβώς τότε ο Καντάφη ετοιμαζόταν να αλλάξει νόμισμα. Ε, τερματίστηκε η δικτατορία, αλλά δεν ακολούθησε δημοκρατία, ε, ακολούθησε αναρχία. Η χώρα τώρα είναι διχοτομημένη και η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη από την εποχή του Καντάφη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφέρον στη χώρα να επανέλθουν κανονικές συνθήκες και να επιστρέψει ομαλότητα αν συνεχιστεί και ο εμφύλιος πόλεμος, αυτό δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης. Ακούσαμε και την Άγγελα Μέρκελ. Ε, Καλή και περισσότερος ακόμα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, ελπίζω πως ε, η ύπατη εκπρόσωπος καταρχήν σύντομα θα αναρρώσει και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το γεγονός πως είστε πάντα πρόθυμος να έρθετε να μας μιλήσετε και στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Μιλάμε σήμερα για τη Λιβύη και πρέπει να σας πω πως με ειλικρίνεια το Σουδάν, η Εμένη, η Λιβύη σήμερα δεν μπορούν να θεωρηθούν πραγματικά κράτη, δεν έχουν κυβέρνηση, δεν έχουμε κάποιον συνομιλητή σοβαρό και αυτό δημιουργεί πολλά από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Γιατί λέει, Λιβύη η κατάσταση είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Έχουμε έθνη, ομάδες, φυλές, ένα νεματηρό και μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος έναν συνομιλητή αξιόπιστο. Η κυβέρνηση της Λιβύης επηρεάζεται από, εξαιρετι... από εξωτερικούς ε, παίκτες, για παράδειγμα την Τουρκία και υπάρχουν ε, στο Τομπρούκ ας πούμε η Αιγύπτη και η Σαουδική Αραβία που επηρεάζουν το παιχνίδι. Ε, δεν μιλάμε λοιπόν για ένα δικτάτορα με τον οποίο θα πρέπει να έρθουμε σε κάποια συμφωνία, αλλά μιλάμε για πάρα πολλές μικρές ομάδες και ξέρω πως ο ΙΕ προσπαθεί να διοργανώσει συνεδριάσεις μεταξύ των διαφόρων, ε, ε, ανάμεσα στις διάφορες φράξεις. Ε, πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν με πιο εμφανή τρόπο αυτή την προσπάθεια που κάνει ο ΟΗΕ, έτσι ώστε να στηθεί μια κυβέρνηση, γιατί έχουμε τις συμφωνίες που υπογράφηκαν τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά για να διαρκέσουν χρειάζεται να παρακολουθούνται μέρα-μέρα και στην Ευρώπη θα πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες που κάνει ο Μπερναρδίνο Λεόν. Και αν θέλουμε να είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές στην Ευρώπη και να δώσουμε μια σταθερότητα στη Λιβύη, θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να συναντηθούν γύρω από το ίδιο τραπέζι όχι μόνο οι τοπικοί ντόπιοι παίκτε, αλλά η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, η ΙΠΑ, γιατί θα πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή και να κλείσει αυτή η τρομακτική κρίση. Κύριε Πρόεδρε, εσείς εδώ Είστε και πρόεδρος απαράλληλα της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης και νομίζω ότι θα πρέπει να επιστρέψει η ειρήνη στη Μεσόγειο και η σταθερότητα. Euh, Ο κύριος Παρνιό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι πολιτικές συζητήσεις ε, που ολοκληρώθηκαν ε, στο Μαρόκο μεταξύ των ε, διαφόρων των μερών και και χαιρετίζουμε το έργο του κύριου Μπερναρντελολεόν. Φτάνουμε τώρα όμως στο πιο λεπτό σημείο της διαπραγμάτευσης και αυτό που απαιτεί ανάληψη ευθυνών ε, από τους μεν και τους δε. Θα πρέπει να πούν ναι ή όχι. Και η κατάσταση είναι κατεπίγουσα. Ε, θα πρέπει ε, να αντιμετωπιστεί η απειλή του ΝΤΑΕΣ που θερίζει στην Λιβύη και πάνω από 100.000 μαχητές ενεργοποιούνται εκεί. Ιδιαίτερα στην παράκτια πόλη της Σύρτα και στην Μισράτα. Είναι πολύ μεγάλος ο δυναμισμός και η παρουσία του Ισλαμικού κράτους στο, στη Λιβύη. Θα πρέπει η χώρα να γίνει κανεί να ελέγξει τα σύνορα και να προστατεύσει την επικράτειά της. Και χαιρετίζουμε τις δηλώσεις ε, της ΥΠΑ της εκπροσώπου ε, για, την, ε, για τα 100 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν αμέσως στην κυβέρνηση που θα αναλάβει στη Λιβύη. Ελπίζουμε να εκτεμευτεί γρήγορα αυτό το κονδύλιο με την ανάληψη τη εξουσίας από τη νέα κυβέρνηση. Ευχαριστώ κύριος Πιοτρόφσκι για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Ε, τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την Αραβική Άνοιξη που οδήγησε και τη Λιβύη στην ανατροπή του Καντάφη, του σταγματάρχη Καντάφη. Και αυτό έγινε με συμμετοχή των ευρωπαϊκών δυνάμεων που εφοδίασαν με όπλα. Ε, βέβαια, με την ανατροπή του Κατάφη ε, δεν αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. Σήμερα έχουμε δύο διαφορετικές πηγές εξουσίας στη Λιβύη και ουσιαστικά κυριαρχεί παντού χάος που το εκμεταλλεύονται το Ισλαμικό κράτος και οι λαθρέμποροι. Και αυτό γίνεται ε, με τη συμμετοχή της Ευρώπης ουσιαστικά και ε, ε πολλές φορές ακόμη και στην αποστολική έδρα είχαμε τρομοκρατικές υπέ, και επιπλέον έχουμε και την προσφυγική κρίση ω συνέπεια αυτού του φαινομένου. Θα πρέπει να συμβάλλουμε στο να σταθεροποιηθεί η κατάσταση εκεί, επί τόπου, στη Λιβύη. Με συνεννόηση με τι ε, Ηνωμένε Πολιτείε και του συμμάχου μα στο ΝΑΤΟ, καθώ και σε συνεργασία με τι χώρε τη Βορειοαφρική. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Φεράν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Η Λιβύη την οποία απελευθέρωσε ο Νικολά Σαρκοζή έχει βυθιστεί στο χάος. Γιατί έκαναν πόλεμο κατά τη Λιβύης η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όντω. δεν μπορεί πια να μας εμποδίζει ο κύριο Καντάφη, ούτε είναι εκεί για να μαρτυρήσει το τι έγινε. Αλλά η απελευθέρωση τη Λιβύη οδήγησε σε Σαριά, Ισλαμικό νόμο, μια ανεργία η οποία έχει ξεπεράσει κάθε, όρο, κάθε ε, όριο, ε, λαθρεμπόριο, ε, ένοπλες δυνάμεις, ε, πολιτοφυλακή και έναν πληθυσμό ο οποίος έχει εκκριζωθεί από τα σπίτια του. Και γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Γιατί στήριξε και προκάλεσε όλα αυτά τα γεγονότα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τεράστιες ευθύνες και στη Συρία και στη Λιβύη και νομίζω ότι τα συμπεράσματα θα πρέπει, στα συμπεράσματα θα πρέπει να καταλήξουμε πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μεγιάν Μιών. Η κατάσταση στη Λιβύη χειροτερεύει συνέχεια. Καθημερινότητα, όπως μας είπε ο Επίτροπος, δυσκολεύει συνέχεια σε αριθμό εκτυπισμένων, σε θύματα και έχουμε τον ΤΑΕΣ, το ISIS, λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών στη χώρα. Παρόλε τι προσπάθειες που έγιναν με τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη για να διευκολύνουμε μια πολιτική λύση, και εδώ πρέπει να τονίσω ποια ήταν η σημαντική προσφορά των Ηνωμένων Εθνών και του ειδικού αποσταλμένου, να σας πω ότι τελικά φτάσαμε σε μια συμφωνία, μια βάση συμφωνία το Σεπτέμβριο που μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο. Πρέπει να δράσουμε, γιατί δεν έχει νόημα ε, να συζητάμε στα λόγια και να καθυστερούμε μια συμφωνία η οποία μπορεί να λειτουργήσει. Θα πρέπει να κλείσουμε με ε, επιτυχία τη διαδικασία που ξεκίνησε στο Μαρόκο. Θα πρέπει να αφήσουμε στους Λίβιους τη δυνατότητα να λάβουν τα ενία του μέλλοντός τους και να επιστρέψουν στην ειρήνη. Και ξέρω πως θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα της τρομοκρατίας ε, και επίσης να καταπολεμήσουν τα διάφορα λαθρεμπόρια τα οποία μαστίζουν τη χώρα. Είναι μια πολύ σημαντική χώρα της Μεσογείου σε ένα γεωγραφικό σημείο που είναι πολύ σημαντικό και γειτονική χώρα. Και ό,τι συμβαίνει εκεί μας επηρεάζει όλους. Αυτό το κενό εξουσία στη χώρα έχει προφανή αποτελέσματα ε, με τα άτομα τα οποία προσπαθούν να διασχίσουν ε, την ε, Μεσόγειο. Η επιχείρηση που θα ξεκινήσει αύριο ελπίζω πως θα προσπαθήσει τουλάχιστον να φρενάρει κάπως τις φρικτές αυτές μαφίες. Και να σας πω πως η κατάσταση είναι εξαιρετική, εξαιρετικά περίπλοκη στο Σαχίλ. Και να σας πω πως όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλες οι γειτονικές χώρες θα πρέπει να σταθούμε επικοδομητικά υπέρ μιας ενωμένης Λιβύης, κυρίαρχης και δημοκρατικής, όπου δεν θα υπάρχει πια βία. Κινδυνεύει η Λιβύη ε, και θέλει σταθερότητα, ενότητα και ειρήνη για να επιβιώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, πάνω από μισό εκατομμύριο ε, άνθρωποι έφτασαν στην Ευρώπη από τη Μεσόγειο. Τρεις χιλιάδες περίπου πνίγηκαν προσπαθώντας να περάσουν τη θάλασσα. Δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό πρόβλημα, είναι και πρόβλημα ασφάλειας. Και πρέπει να σας πω πως η πολύ πρόσφατη ε, πρωτοβουλία για να καταπολεμήσουμε ε, το θέμα αυτό είναι σημαντική, αλλά είναι περίπλοκο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Δεν υπάρχει μια μενωμένη κυβέρνηση και η κατάσταση μάλλον θα χειροτερεύσει κι άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει περισσότερες προσπάθειες ε, σε ένα διαστρωμένο διάλογο και σε μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε ειρήνευση. Οι Λίβοι αξίζουν την ειρήνη και δεν θα πρέπει να είναι όμοιροι μιας μικρής ε, μειονότητας προσπαθεί να κερδίσει με πολεμικά μέσα αυτή, αυτό τον αγώνα. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουν όλοι το εμπάρκο στο εμπόριο όπλων και να στηρίξουν το σχέδιο συμφωνίας που υπάρχει στο τραπέζι. Θα πρέπει εμείς να παραμείνουμε απόλυτα δεσμευμένοι χωρίς να στηρίζουμε τον έναν ή τον άλλον έτσι ώστε να επιληθεί η κρίση, να πετευθεί η κριση να επιτεθει η ειρηνη και να, δημιουργηθεί, να δημιουργηθούν στεναροί κυβερνητικοί θεσμοί. Ευχαριστώ κύριο Σαφχόιζερ. Για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ας ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η τραγωδία στη Λιβύη είναι ο καθρέφτης της ολέθριας εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, υπόδουλος εξωτερικά ε, αμερικανικά συμφέροντα ε, με τον πρόεδρο Σαρκοζή να πρωτοστατεί από τους δόπιους λακέδες. Είναι ένα χάος εκεί των φυλών. η χώρα έχει ε, κοπή Ανατολή-Δύση και από ασφάλεια χάος. Οι ορδές των βαρβάρων του Ισλαμικού κράτους ε, ε, και οι λαθρέμποροι οργιάζουν. Ανθρωπιστικό χάος, 1,5 ε, εκατομμύριο παράνομοι, τσουνάμι λαθρομεταναστών, πολλοί Ισλαμιστές, ε, τρομοκράτες και σήμερα φτάνουν στην Ευρώπη με τη δική σας ολέθρια μεταναστευτική πολιτική. Για να αλλάξει αυτό θα πρέπει να συμφιλειωθούν οι διάφορες φατρίες και να αντιμετωπιστεί το θέμα των παρανόμων επιτόπου. Αλλά αυτό χρειάζεται μια πολιτική άλλη, διαφορετική από τη δική σας που είναι χείριστη πολιτική. Θα πρέπει να επέμπει πάλι η Ρωσία, ίσως και η Αίγυπτος για να αποφύγουμε τα χειρότερα που εσείς μας ετοιμάζετε τώρα. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χαιρετίζουμε με ε, ελπίδα και πολιτική βούληση ε, τη συμφωνία που προσπαθεί να επιτύχει Μπερναδίνο Λεόν, του οποίου η εντολή έληξε την 1η Σεπτεμβρίου. Ε, υπάρχουν πολλοί που προτιμούν το πόλεμο γιατί είναι πιο επικερδής από την ειρήνη σε μια χώρα ε, που σπαράζεται από 40 ε, και πλέον έτη ε, ομής δικτατορίας, φίλιο πόλεμο και σαν να μην έφτανε όλο αυτό ήρθε και το Ισλαμικό κράτος. Γι' αυτό είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο μας να υποστηρίξει και αυτό τη συμφωνία και μάλιστα πριν την 22 Οκτωβρίου που λύγει η εντολή της Βουλής στο Τομπρούκ. Να τεθεί σε ισχύ. Επίση, χρειάζεται χρηματοδότηση για να συνοδευτούν τα πρώτα βήματα και να είμαστε αξιόπιστη. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε ε, σε αυτό το αίτημα για να οικοδομήσουν την ενότητά του οι και να αντιμετωπίσουν τον κοινό εχθρό, το Ισλαμικό κράτος, πριν είναι πολύ αργά. Είναι πάρα πολύ επίγον ε, για να μην πέσει η Λιβύη και ε, η γειτονική την θύμα στα χέρια των τρομοκρατών. Κύριε Επίτροπε, αυτό που χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει επιγόντως και αποτελεσματικά, να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που τώρα ερθώνονται στον ΟΗΕ για τη συμφωνία. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, γνωρίζετε ότι από μια τέτοια κατεστραμμένη χώρα στην νότια όχθη της Μεσογείου θα έχουμε ε, πολύ χειρότερα με αφήξεις ε, ε, διαφόρων μεταναστών προσφύγων στη Βιέννη, στο Καλέ, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο. Ευχαριστώ. Οι διερμηνείς λένε ότι μιλάτε με τέτοια ταχύτητα ορισμένοι που δεν σας προλαβαίνω για να μεταφράζω. Ο κύριος Βάιτεν Χόλτσερ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όταν συζητούμε για τη Λιβύη, συνήθως συζητούμε για τα σφάλματα της Δύσης και όλα αυτά που έγιναν λάθος. Βεβαίως είναι σωστό αυτό, αλλά δεν μας βοηθάει να προχωρήσουμε. Και μάλιστα θα πρέπει να απαντήσουμε γιατί γίνονται όλα τόσο αργά. Επιγόντως θα πρέπει να εξομαλυνθεί εκεί η κατάσταση, δηλαδή να επιτρέψει κρατική υπόσταση, επιστρέψει μάλλον στη Λιβύη. Ε, είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει μια συμφωνία εθνικής ενότητας να αναλάβει τα ενία του κράτους επιτέλους. Ξέρουμε ότι αυτό είναι θέμα του λιβικού λαού, αλλά έχει την ευθύνη της και Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, διότι είναι απαραίτητο. Πρώτον, να υπάρξει σταθερότητα σε αυτή την περιφέρεια που είναι στη γειτονιά μας, Μάρε Νόστρομ είναι η Μεσόγειος, και γιατί αν θέλουμε να αποφύγουμε και τη διεύρυνση ε, του Ισλαμικού κράτου στην Αφρική και τρίτον διότι έχουμε ε, πρόβλημα με τους πρόσφυγες. Μέχρι ένα εκατομμύριο είναι οι άνθρωποι που περιμένουν από εκεί να έρθουν στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ένα λογικό και αξιόπιστο εταίρο για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε τελικά αυτά τα προβλήματα. Η ε, κυρία Ντάλη για ένα λεπτό. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Ανάψτε το μικρόφωνο παρακαλώ κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και αρκετό καιρό ελπίσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για την ειρηνευτική διαδικασία στη Λιβύη. Φτάσαμε στη τελευταία φάση της διαπραγμάτευσης ε, της συμφωνίας ε, που επιβλήθη με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών. Είναι η τελευταία ευκαιρία. Θα πρέπει όμως ε, να μην ε, γίνουμε θύματα αυτών που δεν θέλουν να συνεργαστούν. Θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που θέλουν να συνεργαστούν. Τα Ηνωμένα Έθνη προστατεί σε μια διαδικασία συμφιλίωσης ε, και ειρήνης. Θα πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν τους Λίβιους που θέλουν την πατρίδα τους ελεύθερη, δημοκρατική, χωρίς βία, χωρίς αντιπαραθέσεις, με σταθερότητα και ασφάλεια. Για να συμβούν όμως όλα αυτά είναι απαραίτητο όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν δραστήριο ρόλο στη διαδικασία σταθεροποίηση αυτή τη χώρα. Ευελπιστούμε ότι θα συναθεί τελικά η Ειρηνευτική Συμφωνία, θα εφαρμοστεί και εμπράκτο και θα χαράξει το δρόμο για μια σταθερότερη και ασφαλέστερη Λιβύη. Η κυρία Κριστέα, για ένα λεπτό. Ο κύριο Κριστέα, συγγνώμη, για ένα λεπτό. Τέσσερα χρόνια μετά από τη στιγμή που κατέβηκαν στους δρόμους για να τήσουν αξιοπρέπεια, δημοκρατία, ελευθερία, οι Λίβοι ζουν σε μια χώρα διαιρεμένη, βίαιη η κρίση έχει επηρεάσει και τον άμαχο πληθυσμό που υποφέρει με εκτοπισμένους και με μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση που εξαπλώνεται. Σήμερα χρειάζεται να δείξουμε ευθύνη και να δείξουμε θάρρος. Η τελευταία συμφωνία την οποία διαπραγματευόμαστε είναι η τελευταία ευκαιρία και θα πρέπει έτσι να έχουμε μια βιώσιμη λύση για τη χώρα. Εξαρτάται από τα εμπλεκόμενα μέρη να αποδείξουν πως πραγματικά είναι δεσμευμένοι υπέρ μιας δημοκρατικής νέας Λιβύης που θα προσφέρει σταθερότητα, ειρήνη και ευημερία στους Λίβιους που τους αξίζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ό,τι μπορεί για να στηρίξει ε, αυτή τη συμφωνία, αλλά θα πρέπει τα όσοι διαπραγματεύονται τη συμφωνία να βρουν μια συμφωνία που θα φέρει πραγματική ειρήνη. Ο κύριος Φρόιντ είναι ο επόμενος μιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα πιο πρόσφατα νέα από τη Λιβύη είναι απογοητευτικά. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν δεν έχει γίνει κάτι αποφασιστικό, το παράδειγμα Λιβύη δείχνει τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν συνεννοείται με τα Ηνωμένα Έθνη και κινητοποιεί τις διπλωματικές δυνάμεις. Αυτή η Στη βαρύ όμως εξωτερική πολιτική δεν είναι απαραίτητη αποκλειστικά απέναντι στη Λιβύη αλλά και σε άλλες αιστείες ανάφλεξης θα πρέπει να είμαστε παρόντες περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα. Σε ό,τι αφορά τη Λιβύη θα πρέπει να πούμε στους ηθήνοντες ε, ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση προς την ειρήνη. Θα πρέπει τα αντιμαχόμενα μέρη να καταλάβουν ότι αυτή η ευκαιρία που έχει τώρα ε, η χώρα είναι μια ευκαιρία που δεν πρόκειται να ξανάρθει τόσο γρήγορα. Και αν παραταθεί ο φίλος πόλεμος, αυτό σημαίνει ε, πρόβλημα για την δική μας ασφάλεια ενδεχομένως και για την κοινωνική μας συνοχή με το προσφυγικό. Ευχαριστώ. Μπένι και εσείς ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Βρισκόμαστε σε μια πολύ αποφασιστική και κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Λιβύης. Αυτή τη στιγμή οι εμπλεκόμενοι ίσως καταλήξουν συμφωνία για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας χάρη στην προσπάθεια του Μπερναρντίνο Λεόν με την υποστήριξη της ύπατης εκπροσώπου Μογκερίνη. Ολόκληρος ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια του στη Λιβύη και περιμένει ε, να δει αν οι εκπρόσωποι του Τομπρού και της Τρίπολης έχουν βούληση να καταλήξουν συμφωνία. Βέβαια, τα νέα που ακούμε είναι σχετικά αποθαρρυντικά, όπως μας είπε η κυρία, η Γκόμες. Πολλά εκκρεμή προβλήματα υπάρχουν. εκπροσώπευση των εμπλεκομένων, εφαρμογή της συμφωνίας, ανάγκη διαμόρφωσης μια ζώνης ασφαλείας, προκειμένου να παρεμποδιστούν οι λαθρέμποροι και οι μαφίες κάθε είδους να εφαρμόσουν το έργο τους. Επίσης θα πρέπει πάση θυσία να επανέλθει η ειρήνη στη Λιβύη. Αυτό όμω είναι ένα θέμα που βρίσκεται στα χέρια των ίδιων των Λιβύων. Θα ήταν κρίμα να διαλυθεί περαιτέρω η Λιβύη, θα έχει καταστραφικές συνέπειες για την Ευρώπη. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνή κοινότητα θέλουν να πετύχουν, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι ξέρουμε ποια είναι τα διδάγματα του παρελθόντο. Γιατί για μια φορά ακόμα μετά τη σύρρηξη αποτυγχάνουμε. Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Γιατί 800 εκατομμύρια δώσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Και αυτά ε, το θυμόμαστε. Έχουμε ε, ε ευθύνε. Αλλά τι θα γίνει με αυτέ τι ομάδε οι οποίε δεν σέβονται τα ανθρώπινα και τα δημοκρατικά δικαιώματα. Ένα νέο καντάφι βάλουμε στη θέση του προηγούμενου. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πως δεν ε, θα επιτρέψουμε στις δυνάμεις της καταστροφής να υπερισχύσουν. Χρειαζόμαστε μια ειρηνική συμφιλίωση υπέρ του λιβικού λαού, όχι μόνο μέσω ε, των φυλακών που δημιουργούμε ελέγχοντας τη μετανάστευση προς τις ακτές μας. Χρειαζόμαστε να εξασφαλίσουμε το μέλλον για τις χώρες αυτές ε, και να εξασφαλίσουμε και τα νότια και τα θαλάσσια σύνορα της χώρες αυτής και να μην επιτρέπουμε ομάδες να προσελκύονται στο ISIS λόγω της κατάστασης. Η αποτυχία της δημοκρατικής μετάβασης στην Λιβύη οδήγησε στη δημιουργία ενός καυτού σημείου της τρομοκρατίας. Και εμείς πρέπει να κατεβάσουμε λίγο τη θερμοκρασία στη Λιβύη για να είναι πιο ασφαλής και για τους ίδιους κατοίκους. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε τώρα να μπούμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχω τη δυνατότητα να δώσω μία παρέμβαση σε κάθε πολιτική ομάδα. Αυτό επιτρέπει ο χρόνος, ανάλογα με τα δικά σας αιτήματα. Ο κύριος Σογκορίνο, πρώτος για ένα λεπτό. Thank Σας ευχαριστώ. Τέσσερα χρόνια μετά την ανατροπή του Καντάφη, η Λιβύη υποφέρει από μια καταστροφική κατάσταση με οικονομικές, ανθρωπιστικές και πολλές άλλες διαστάσεις. Τώρα βρισκόμαστε στα πρόθυρα μια σύναψη συμφωνία μεταξύ των δύο φατριών, προκειμένου να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση εθνική ενότητα. Έτσι θα μπορέσουμε να περάσουμε σε μια δεύτερη φάση στη Λιβύη και να καταφέρουμε και εμείς πιο αποτελεσματικά να εμποδίσουμε τους διακινητές στα διεθνή χωρικά ύδατα. Όσο μένει αποσταθεροποιημένη η Λιβύη, οι πολέμαρχοι και οι μαφιόζοι θα υποφελούνται από το χάος και θα οδηγήσουν στην εξαθλίωση και στην έξοδο από τη χώρα πολλές ακόμη χιλιάδες Λιβύων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίτσι. Όχι. Φρουντζούλικα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι είμαι τυχερός. Πιστεύω ότι είναι και, καινή ώρα να κάνουμε ένα παφησιστικό βήμα και να φτιάξουμε ένα δημοκρατικό κράτο στη Λιβύη και μια κυβέρνηση εθνική ενότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκε και οι προσδοκίε του λιβυκού λαού. Ολόκληρη η περιοχή υφίσταται την αποσταθεροποίηση τη τρομοκρατία. Θα πρέπει λοιπόν να κοινού με τη διεθνή κοινότητα να θέσουμε ένα τέρμα στην αντιπαράθεση και να επαναφέρουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα. Η αποτελεσματική πολυμέρεια στο παρελθόν έδειξε ότι οι διεθνεί κρίσει μπορούν να επιληθούν αν όλε οι εμπλεκόμενε πλευρέ είναι πρόθυμε να επανέλθουν στο διάλογο και σε συνεργασία με διεθνεί παράγοντε να εφαρμόσουν και εμπράκτω τη συμφωνία. Θα πρέπει να επαναφέρουμε την ασφάλεια στη Λιβύη. Έτσι θα μειωθεί ο αριθμό των προσφύγων προ την Ευρώπη και θα χαλαρώσει και η πίεση προ τα εξωτερικά μα σύνορα για να μπορέσουν οι μετανάστε να μείνουν στη χώρα του. Γι' αυτό όμω χρειάζονται σταθερή Λιβύη και ε, εξασφάλιση των δημοκρατικών του δικαιωμάτων. Σα ευχαριστώ και ευχαριστώ που τηρήσατε και τον χρόνο. Κύριο Μαριά, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στη Λιβύη αναδεικνύει τι νέε προκλήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο προσφυγικό έχουμε πάνω από τετρακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες που προσπαθούν να διαφύγουν από τον εμφύλιο πόλεμο και έρχονται στην ευρώπη. το ερώτημα που υπάρχει είναι ποιοι ενισχύουν τους τζιχαντιστές αυτή τη στιγμή στην ε, λιβύη όπως και στη συρία ποιος είναι ο ρόλος της τουρκίας ποιος είναι ο ρόλος άλλων δυνάμεων. γνωρίζει η κομισιόν ότι σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες το πλοίο χαντάντ ένα το οποίο έφυγε από την αλεξανδρέτα με στόχο να πάει στη λιβύη σε περιοχή στη μισράτα εκεί που υπάρχουν οι τζιχαντιστές συνελήφθη έξω από την κρήτη με παράνομο οπλισμό πέντε όπλα 500.000 σφαίρες. έχετε εικόνα στην κομισιόν πού πήγαιναν αυτά τα όπλα τα οποία έφυγαν από λιμάνι της τουρκίας; τι γίνεται με τον παράνομο οπλισμό στα ζητήματα αυτά; ποιος εξοπλίζει πλέον τους τζιχαντιστές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κιουτσούκ, παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. στην Λιβύη οι αντιμαχόμενες δυνάμεις ουσιαστικά προκαλούν ε, τα πάνδυνα στον άμαχο πληθυσμό. Τώρα έχουμε τον ειδικό επεσταλμένο Μπερναρντίνο Λεόν και τις προσπάθειες του να χαράξει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τη Λιβύη. Βέβαια δεν είναι τέλεια η συμφωνία, αλλά δυστυχώς ε, οι δύο κυβερνήσεις στη Λιβύη δεν δίνουν καν ε, οποιαδήποτε, δεν δείχνουν οποιαδήποτε σημάδι, οποιαδήποτε βούληση ε, σύναψη συμφωνία και ανέβρεση μια λύση. Η κυρία Μογκερίνη θα πρέπει να συνεχίσει τι προσπάθειε εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να επαναφέρει τι αντιμαχόμενε πλευρέ στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, προκειμένου να συσταθεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας και συμφιλίωσης. Γιατί αν αποτύχουμε σε αυτή την προσπάθεια, αφήνουμε ουσιαστικά ανοιχτή την πόρτα για περαιτέρω προσφυγικά ρεύματα. Κύριε Κονέτσνα, για ένα λεπτό κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολλοί πρόσφυγες που ε, πέφτουν στη θάλασσα, στη Μεσόγειο, για να ξεφύγουν από την κατάσταση αυτή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και έχει τραγική κατάληξη πολλές φορές. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να καταβάλουμε όλες τις πολιτικές ε, προσπάθειες για να βοηθήσουμε τη Λιβύη να σταθεί στα πόδια της, να έχει θεσμούς που να βάλουν τάξη στη χώρα αυτή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλα κράτη του ΝΑΤΟ ε, αναμίχθηκαν στις κρατικές δομές της χώρας αυτής σήμερα έχει καταρρεύσει. Χρειάζεται ανοικοδόμηση, μεταπολεμική. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση. Δεν πρόκειται να επανέλθει σταθερότητα στη χώρα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να δούμε σε ποια κατάσταση, η κτρή κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε τώρα να λαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Η κυρία Ντότς. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μα δώσετε κάποιε λεπτομέρειε για τη βοήθεια που θα χορηγήσουμε στη Λιβύη και επιπλέον 100 εκατομμύρια ε, ένα συμπληρωματικό ποσό στα υπάρχοντα ήδη προγράμματα. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι αυτή η γενοδορία, αν υλοποιηθεί, θα συνδυαστεί με εχέγγυα και εγγύηση που θα πρέπει να δώσει η Λιβύη για ελευθερία, για ε, ανεξιθρησκεία και για σταμάτημα των διωγμών των θρησκευτικών μειονοτήτων. Επί Καντάφη, οι, οι, οι τρομοκράτες του Ήρα που ήταν υπεύθυνοι για πολλές ενέργειες και θύματα στη Βόρεια Ιρλανδία συνέχισαν τη δράση τους και μάλιστα στο Westminster στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε ότι ε, ε ένα τμήμα των ε, παγωμένων ε, περιουσιακών στοιχείων της Λιβύης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποζημίωση των θυμάτων του Ήρα γιατί κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην κοινοτική νομοθεσία. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Ε, και αν ε, όχι, μπορείτε να συνεργαστείτε με τα θύματα των τρομοκρατών του Ήρα ώστε να προωθηθούν κάποιες ενέργειες αποζημίωσης και να διορθωθεί αυτό το τεράστιο κακό που κατέφερε ο Ήρα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο Επίτροπος ο κ. Στυλιανίδης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο πλούσια αυτή συζήτηση και για την τόσο ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων που θα διαβιβάσω φυσικά στην ύπατη εκπρόσωπο. Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών τις επόμενες εβδομάδες και βεβαίως ελπίζουμε να επιτευχθεί συμφωνία και να υπογραφεί από όλα τα ενεχόμενα μέρη τις ερχόμενες μέρες. Είμαστε αισιόδοξοι ότι ε, το αναγνωρίζουν αυτό και καταλαβαίνουν όλα τα ενεχόμενα μέρη ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Έχει έρθει η ώρα να ε, σκεφτούμε το μέλλον της Λιβύης. Η η οικονομία της χώρας έχει καταρρεύσει και έχει καταστραφεί επίσης και ο κοινωνικός ιστός της. Εμείς είμαστε έτοιμοι να επιβάλλουμε κυρώσεις σε εκείνους που το τελευταίο έτος απέδειξαν ότι είχαν στόχο να υπονομεύσουν τις συνομιλίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να δεχτεί διχοτόμηση της Λιβύης η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να δεχθεί νίκη οποιασδήποτε πλευράς η οποία θα επιβάλλει ε, το δικό της νόμο με τη βία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να δεχθεί ε, ότι δεν θα υπάρχουν ε, ελεύθερες δομές ανεξάρτητες όπως είναι ε, οι ε, αναπτυξιακοί οργανισμοί, οι εταιρείε πετρελαίου. Ε, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι δεν θα είναι ουδέτερες αυτές οι δομές και ότι θα συμμετέχουν στη μία την άλλη πλευρά. Η ουδετερότητα ήταν εκείνη που έχει διατηρήσει τη χώρα ενωμένη και μόνο έτσι θα μπορέσει να διατηρηθεί και στο μέλλον. Νομίζω ότι αυτή είναι δική μας ηθική ευθύνη και χρέος ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πρόεδρο, ευχαριστούμε τον Επίτροπο κύριο Στυλιανίδη και θα σας πω ότι